we um, Καλησπέρα, συνάδελφοι. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσει, εγκρίνεται η ημερήσια διάταξη. Σήμερα δεν έχουμε δανέζικα, μαλτέζικα, κροατικά και ιρλανδικά και 6,5 ώρα έχουμε ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ετοιμάστε τις κάρτε σα και τέλο στις ανακοινώσεις ε, του Προέδρου έχουμε έγκριση ε, πρακτικών ε, των συνεδριάσεων 9 έως 12 Απριλίου. Δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, εγκρίνονται. Περνάμε λοιπόν τώρα στο μόνο θέμα της ημερησίας διάταξης πέρα από την ψηφοφορία που είναι η παρουσίαση από τον Επίτροπο τον κύριο Κίνγκ το του θέματος της Ένωση Ασφαλείας. Και να σα ευχαριστήσω εδώ πέρα για την προπαρασκευαστική συνεδρίαση της 5 η Δεκεμβρίου με την Europol και τις σχετικές ε, μονάδες ε, του άρθρου 19. Νομίζω ότι ήταν εξαιρετική προετοιμασία για τη σημερινή μας ε, συνεδρίαση και γνωρίζω βεβαίως πως θα έρθουν και άλλοι συνάδελφοι σιγά σιγά αλλά νομίζω είναι πολύ σημαντικό να έχουμε αυτή την συνάντηση όπως, έτσι, όπως αποφάσισαν οι συντονιστές να εστιάσουμε δηλαδή δύο φορές το χρόνο σε ένα συγκεκριμένο θέμα με τον Επιτροπό. Θα θυμάστε ότι η πρώτη έγινε στις 23 Μαΐου και εστίασε στην εφαρμογή και στην χρήση υφιστάμενων πληροφοριών και σήμερα θα δούμε την αντιμετώπιση των τρομοκρατικών αφηγημάτων. Όπως είπα λοιπόν, έχουμε... Είχαμε την προπαρασκευαστική συνεδρία στις 5 Δεκεμβρίου και σήμερα θέλουμε να ακούσουμε από τον Επίτροπο ποια είναι η άποψή του και η ανάλυση του για τις ε, κυρίες αυτές προσεγγίσεις και το πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την νομοκρατική προπαγάνδα και είδαμε νομίζω τα είδαν και οι συνάδελφοι για την διατάραξη, το κατέβασμα τέτοιου περιεχομένου, η ανακατεύθυνση, καμπάνιες και σχεδιασμός του μηνύματος και για, συγχρονισμός, και για συγχρονισμό των μηνυμάτων των κυβερνήσεων και είχαμε και ένα πάρα πολύ καλό έγγραφο του Κοινοβουλίου που παρουσιάζει την σχετική έρευνα. Και παρακαλώ να το δείτε εάν δεν το έχετε δει. Να ρίξετε μια ματιά. Οπότε, γνωρίζουμε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει έναν εθελοντικό κώδικα συμπεριφοράς για το κατέβασμα παράνομου περιεχομένου μέσω της μονάδας ε, παραπομπής διαδικτύου της Europol αλλά βεβαίως η σαφήνεια και η έλλειψη κοινών ορισμών επίσης ήταν κάτι το οποίο συζητήσαν οι συναδελφοί την Τετάρτη που μας πέρασε. Έχουμε λοιπόν ένα βασικό ζήτημα εδώ για την εξαμενία συνάντησή μας. Χαίρομαι που είναι εδώ ο Επίτροπος και ήρθαν και οι βουλευτές. Κύριε Επίτροπε, να σας δώσω τον λόγο για 10 λεπτά. Ε, να πω επίσης πως ε, συνάδελφοι ε, επίσης ε, και από την Επιτροπή περί τρομοκρατίας βρίσκονται εδώ σήμερα. Λοιπόν, έχετε τον λόγο για 10 λεπτά κύριε Επιτροπέ και μετά θα δώσω τον λόγο στους ε, συναδέλφους. Ευχαριστώ που με καλέσατε για το διάλογο για την ασφάλεια. Έγινε πολύ μεγάλη προετοιμασία για το θέμα αυτό. Ίσως δεν θα καλύψω όλα, αλλά ίσως στις ερωτήσεις και απαντήσεις να καλύψουμε τα κενά. Θα είμαι κάπως πιο γενικός, αν επιτρέπετε, να δούμε τι κάνουμε για την πρόληψη. Δοθέτω ότι προφανώς η πρόληψη είναι καλύτερη από τη θεραπεία. Θα αναφερθώ στη χρηματοδότηση των τρομοκρατών και πώς μπορούμε να τους αποκόψουμε από τους οικονομικούς πόρους, αλλά αφού με καλέσατε θα εστιαστώ με το πώς θα αντιμετωπίσουμε τον εντοπισμό της ριζοσπαστικοποίησης, να δούμε κάποια σημάδια που μπορούν να μας ειδοποιήσουν γι' αυτό, πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο που πλήττει ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και ανθρώπους. Και πρέπει να δούμε και το χώρο στον οποίο κινούνται οι τρομοκράτες. Όσο το εξετάζουμε αυτό, βλέπουμε ότι πρέπει να βρούμε τα ριζικά αίτια. Ριζοσπαστικοποίηση προς κάποια ιδεολογία τρομοκρατική, και θα πρέπει να αυξήσουμε τις αντοχές των ατόμων, των κοινοτήτων κατά της προπαγάνδας και της ριζοσπαστικοποίησης. Το διαδίκτυο παίζει σημαντικό ρόλο στις επιθέσεις που έχουμε δει να πραγματοποιούνται τους τελευταίους μήνες. Χρησιμοποιούνται όλοι οι τρόποι για να προετοιμάσουν τα άτομα για να πραγματοποιήσουν τις επιθέσεις και να τους παρακινήσουν να επιτεθούν και να διαδώσουν προπαγάνδα. Λοιπόν, η προπαγάνδα και τα εγκλήματα γίνονται και στο διαδίκτυο και εκτός διαδικτύου και πρέπει όλες τις στοιχείες να τις λαμβάνουμε υπόψη α, σοβαρά. Κανένα φορέας μόνο του δεν μπορεί να πετύχει το στόχο της αντιμετωπίσης τρομοκρατίας. Το είδατε και από αυτά που μας είπαν μάρτυρες πρόσφατα. Η κυβέρνηση, η κοινωνία των πολιτών, ε, οι πολίτες πρέπει να συνεργαστούν. Το διαδίκτυο του το Internet Forum της Ευρωπαϊκής Ενώσεως προσπαθεί με τη συμμετοχή διαφόρων ειδικών και με διάφορου φορεί και διάφορε κόμβου επικοινωνία Ευρωπαϊκή Ενώσεω, με συμμετοχή πανεπιστημιακών, με ενδιαφερομένου για το θέμα. Όλοι προσπαθούν να κινηθούν για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα μαζί με εταιρείε. Είναι αυτό το Internet Forum για να συζητήσουμε αυτά τα προβλήματα. Τα τελευταία δύο χρόνια αυτό κάναμε. Έχει κάνει πολύ καλή δουλειά το δίκτυο αυτό, αντιμετωπίζοντας την προπαγάνδα αλλά και υποστηρίζοντας και διάφορα εναλλακτικά αφηγήματα. Τελευταία εβδομάδα είχαμε την τρίτη ετήσια διπουργική συνεδρίαση στις ε, Βρυξέλλες. Στο τέλος της ε, συνεδριάσεως ο Δημήτρης Αβραμόπουλος και υποφανόμενος και εμείς θεωρήσαμε ότι κινούμεθα προς αυτή κατεύθυνση. Πολύ σημαντικές εταιρείες χρησιμοποιούνται συστήματα αυτόματου εντοπισμού για να ελέγχουν βίντεο αναρτήσεις λογαριασμού στο Twitter, στο YouTube, στο Facebook ε, που επίσης ε, διαδίδουν προπαγάνδα. Και επίσης υπάρχει και ένα κέντρο που συγκεντρώνει τις πληροφορίες βάσει δεδομένων που περιέχει 40.000 στοιχεία ώστε αν κάτι αναρτηθεί κάπου να μην μπορεί να αναρτηθεί κάπου αλλού, εντοπίζεται αυτό το σύστημα. Επίσης στο Europol γίνεται έξοχη δουλειά πάνω από 40.000 ε, αναρτήσεις παρέπεμψαν αλλά έχουν να αντιμετωπίσουν 100 διαφορετικές πλατφόρμες. Όχι μόνο στις μεγάλες πλατφόρμες για αναρτήσεις και μηνύματα, αλλά και μικρότερες πλατφόρμες. Τα κράτη-μέλη παίρνουν το θέμα σοβαρά, κάτι που ελπίζαμε, και προσπαθούν να δουν τι δυνατότητες έχουν, ώστε να εντοπίζουν και να παραπέμπουν περιεχόμενο ή να κατεβάζουν το περιεχόμενο. Δεν τελειώσαμε ακόμα, καλά τα πάμε, αλλά πρέπει να πάμε καλύτερα Πρέπει να επιταχύνουμε το έργο μας, ε, πρέπει να παρακολουθούμε αυτά που κάνουμε, ώστε να έχουμε συνέπεια στην αντιμετώπιση, να επικρατεί διαφάνεια. Δεν έχουμε συγκεκριμένα ε, στοιχεία ή ταχύτητα ε, διαγραφής αυτών των μηνυμάτων, παρόλο που όλοι θέλουν μέσα σε μία ώρα το πολύ, τη χρυσή ώρα να κατεβαίνουν και στην, άση, στην βάση δεδομένων πρέπει να δούμε πόσο γρήγορα μπορούμε να εντοπίζουμε περιεχόμενο και να το διαγράφουμε καμιά φορά πρέπει να δούμε πώς διαδίδονται οι πληροφορίες και με τους διαφόρους δυνάμεις ασφαλείας. Ε, έχουμε ακόμα μικρομεσές εταιρείες οι οποίες δεν συμμετέχουν πλήρως σε αυτή την προσπάθεια και εκείνοι που αναρτούν την προπαγάνδα προσπαθούν να βρούνε τον αδύναμο κρίκο. Αν κάποια πλατφόρμα κατεβάσει τα μηνύματά τους πάνε σε άλλη. Πρέπει να δούμε τι κάνουμε αυτό το, τι γίνεται με το οικοσύστημα αυτών των πλατφορμών. Θέλουμε όλη αυτή τη δουλειά να την κάνουμε επί εθελουσίας βάσεως. Επ' αυτής της βάση έχουμε σημειώσει πρόοδο, αλλά όπως είπε και ο πρόεδρος Γιούνκερ στην επιστολή του που απέφθηνα στο Κοινοβούλιο, παρακολουθούμε την πρόοδο, εξελογούμε κατά πόσο συμπληρωματικά μέτρα απαιτούνται, ούτω ώστε να εξασφαλίζουμε ταχεία και πρακτική αντιμετώπιση του φαινόμενου. Εντοπίζουμε και να κατεβάζουμε το ε, τα μηνύματα από το διαδίκτυο και να αλλάξουμε ενδεχομένως και το ρυθμιστικό και νομοθετικό πλαίσιο. Και μετά πρέπει να κάνουμε και αντιπροπαγάνδα, το αντιαφήγημα για να αντιμετωπίσουμε τις ρίζες της βίας και της πρακτικοποίησης και να δούμε όμως πώς μπορούμε να αλλάξουμε την εικόνα που απευθύνουν τα μηνύματα αυτά προς τους ανθρώπους. Έχει θετικό ρόλο να παίξει το διαδίκτυο να μπορούμε να πλησιάσουμε τους απογοητευμένους, τους πικραμένους. Ε, το συζητήσαμε αυτό και στο Internet Forum την περασμένη εβδομάδα και συζητήσαμε και την έξοχη δουλειά που έχει γίνει για να προσπαθήσουμε να δώσουμε την δυνατότητα στην κοινωνία των πολιτών να βοηθήσει στην προσπάθεια. Όπως ξέρετε έχουμε σοβαρά προγράμματα πάνω από 10 εκατομμύρια, μάλλον μέχρι 10 εκατομμύρια ευρώ έχουμε διαθέσει σε 10 φάσεις να συμπληρώσουμε τις εθνικές προσπάθειες και τις προσπάθειες που υποστηρίζονται από τις εταιρείε του διαδικτύου τις ίδιες. Ε, στην πρώτη φάση έχουμε το κέντρο αριστείας που προσπαθεί να καταρτήσει την κοινωνία των πολιτών. Πάνω από 250 οργανώσεις έχουν συμμετάσχει σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξεκινήσαμε διαγωνισμό και καλούμε την κοινωνία των πολιτών να ζητήσει χρηματοδότηση για 6 εκατομμύρια ευρώ για διάφορα προγράμματα για να αντιμετωπίσουν την προπαγάνδα, τη βία στο, ε, διαδίκτυο με αντίθετα μηνύματα. Έτσι απηχούμε πολλές από τις συστάσεις που έχουν προέρθει την Επιτροπή σας ε, και ε, από επαφές που είχαμε δεν θα είναι μεμονωμένες εκστρατείες, πρέπει να ενταχθούν σε μια ενιαία στρατηγική επικοινωνίας ε, για δράση, για να καλύψουμε τα κενά και οι διαδραστικές αυτές ε, πρωτοβουλίες θα πρέπει να τύχουν υποστηρίξεως και εκτός διαδικτύου, θα πρέπει να δούμε ποιος είναι ο στόχος, ποιο είναι το ακροατήριο οι δράσεις μας να φτάνουν στους ευάλωτους, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να καθορίσουν προσμετρήσιμους συγκεκριμένους στόχους που μετά θα αξιολογηθούν. Επίσης θέλουμε να βελτιώσουμε την αντίληψή μας για τη βία ριζοστικοποίηση, ούτως ώστε να είναι σε καλύτερη θέση ε, τα μέτρα μας να αντιμετωπίσουν αυτά τα προγράμματα ε, θα πρέπει να έχουμε επιστημονικά εργαλεία που καταλήγουν σε προτάσεις ε, για διαμόρφωση πολιτικής ε, και εμπειρογνώμονες για τη ριζοσφαστικοποίηση. Διάφορα προγράμματα βασίζονται στον εντοπισμό τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο και χρηματοδοτήσαμε περίπου 15 τέτοια προγράμματα πρόσφατα. Δώσαμε περίπου 13 εκατομμύρια ευρώ Λοιπόν, έχουμε το δίκτυο και το κέντρο αριστεία για τη ριζοσπαστικοποίηση και βοηθά τι κοινωνικέ ομάδε να ανταλλάξουν ιδέε και να μάθουν οι μένα του δέου, οι δραστηριοποιούνται εκεί. Τα κράτη-μέλη αυξάνουν τι υποδομέ, του πόρου και τι δυνατότητε που έχουν και απαιτούνται για να υπάρχει καλή επικοινωνία και εξαρτή επικοινωνία από τι δημόσιε αρχέ και από την κοινωνία των πολιτών και από άλλε αξιόπιστε φινέ. Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Στρατηγικών Επικοινωνιών που ξέρω ότι εξετάσατε βοηθά τα κράτη-μέλη να αναπτύξουν δικέ του στρατηγικέ και απαντήσει σε αυτά τα θέματα αυτά. Όλη αυτή η δουλειά νομίζω ότι είναι σημαντική αλλά συμφωνώ με την άποψη που εκφράσατε στην έκθεσή σας που αναφέρατε και στις ότι η στρατηγική επικοινωνία θα πρέπει να παραμείνει στο κέντρο τη αντιτροκομοκρατική μα πολιτική. Πρόσφατα Δημιουργήσουμε την ομάδα υψηλού επίπεδου για τη ζωσπαστικοποίηση με τη συμμετοχή Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κρατών Μελών, ακαδημαϊκών, ερευνητών, αρμοδίων του τομέα, όλων όσων κινούνται σε αυτόν τον τομέα, ώστε να συναθρήσουμε εκείνους που είναι στην πρώτη γραμμή μέσω παιδείας, με συμμετοχή τους σε κοινωνικά δρόμενα και την τοπική αυτοδιοίκηση, ούτως ώστε από κοινού να έχουμε τα σωστά αποτελέσματα η πρώτη διάμεσα έκθεση παρουσιάστηκε την περασμένη εβδομάδα. Ζητεί την αύξηση κατά πολεμήσεω τρομοκρατική προπαγάνδα. Υπογραμμίζει τη σημασία οι φυστάμενοι φορεί που ασχολούνται με αυτόν τον τομέα να κινούνται ακόμα. Ζητά πιο στεναρή διαθρωμένη απάντηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα προσπαθήσουμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ενώσεω για να βοηθήσουμε να υποστηρίξουμε τι αρχέ των κρατών μελών και την κοινωνία των πολιτών να κάνουν το έργο του αποτελεσματικά. Κλείνοντα, διότι έχω μερικά δευτερόλεπτα που μένουν, αλλά παρακαλώ να είστε υπομονετικοί απέναντί μου και να καταλήξω με κάποια λόγια για τη χρηματοδότηση των δημοκρατών. Ξέρω ότι αυτό είναι ένα θέμα που αφορά την Επιτροπή σα. Όλοι κατανοούμε τη σημασία του έργου που κάνουμε. Ε, νομίζω ότι κάναμε κάποια πρόοδο. Πρέπει να πω ότι θα ήταν υπέροχο αν θα μπορούσαμε να ολοκληρώσουμε τι εργασίε μα στην ε, πέμπτη αναθεώρηση της οδηγίας για το ξέπλυμα του παράνομου χρήματο. Ε, ο κύριο Κάρεν και η κυρία Σαρτζεντίνη έχουν εργαστεί άοκνα επ' αυτού. Ελπίζουμε να, ελπίζαμε να ολοκληρωθεί η επιστονική παιδεία. Εμεί θέλουμε να σημειώσουμε πρόοδο και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Ξέρουμε γιατί η διαφάνεια τη πραγματική ιδιοκτησία και τη πληροφορία είναι πάρα πολύ κρίσιμη σημασία και θα πρέπει να υπάρχει και η διαφάνεια για τα καταπιστεύματα. Λοιπόν, ένα, κέντρο, ένα κεντρικό αρχείο τραπεζικών λογαριασμών θα βοηθούσε στο να καταπολεμήσουμε τη χρηματοδότηση των δημοκρατών. Ελπίζω στον επόμενο τριμερή διάλογο να βρούμε λύση. Εδώ και ένα χρόνο προτείνω μια οδηγία για την αρμόνιση του ορισμού των ποινικών κυρώσεων για το ξέπλυμα χρήματο, συμπληρώνοντα την οδηγία τη σχετική για την καταπολέμηση του φαινομένου αυτού και θα βοηθούσαμε έτσι τη συνοριακή συνεργασία. Και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα ψηφίσετε αργότερα σήμερα το απόγευμα, σήμερα το βράδυ πάνω σε αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη δουλειά που κάνετε πάνω σε αυτό. Θα ήθελα να καλωσορίσω τη θετική ψηφοφορία την περασμένη εβδομάδα στην κοινή συνεδρίαση που είχατε για την πρόταση για την ενίσχυση των ελέγχων για, το μετρητό, για τα μετρητά που κινούνται δυσυνοριακά εκτός Ευρωπαϊκής Ενώσης. Ευχαριστώ όλους όσους το επεξεργαστήκατε αυτό. Το τρίτο θέμα ήταν να διευκολύνουμε αμοιβαία αναγνώριση του παγώματο στοιχείων ενεργητικού και κατασχέσεων ε, λογαριασμών και προσιακών στοιχείων σε ποινικέ υποθέσει. Υποστηρίζω ένθερμα το έργο τη Greensberg ε, της κυρίας Γκρινσμπερκ που έκανε σε αυτό το θέμα. Ε, ελπίζω όλα αυτά να ολοκληρωθούν μέχρι το επόμενο καλοκαίρι. Γιατί τα αναφέρω αυτό, διότι πέρα από το πρόσφατο πακέτο για την κυβερνοασφάλεια που συζητήσαμε προηγουμένω, επίση κάναμε και μια πρόταση για την κατονέμηση τη απάτη και την ε, παραχάραξη μη μεθόδων πληρωμή μη πλην μετρητών. Αυτό συμπληρώνει ήδη το επιτελεστέν έργο και το επιτελούμενο έργο και ετοιμάζουμε μία πρόταση. Πρόταση οδηγία, ούτω ώστε οι αρχέ επιβολή του νόμου έχουν πρόσβαση στο εθνικά μητρώα ε, τραπεζικών λογαριασμών που θα δημιουργηθούν, ούτω ώστε να μπορούν οι αστυνομικέ αρχέ και άλλε αρμόδιε αρχέ να έχουν πρόσβαση σε τραπεζικού λογαριασμού και να υπάρχουν ανταλλαγέ πληροφοριών με ομολόγου σε άλλα κράτη-μέλη βάσει των ισιών των κανόνων. Επισχυράζομαστε πρωτοβουλίε για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των διαφόρων κέντρων πληροφοριών για οικονομικά θέματα, καταπολεμής οικονομικού εγκλήματος και θα δούμε πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε αναλογικά συμπληρωματικά μέτρα για να υποστηρίξουμε το έργο που κάνετε και εσείς όσον αφορά την αντιμετώπιση της χρηματοδοτής των τρομοκρατών. Τέλος, αύριο στο Κολέγιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εγώ μαζί με τον Δημήτρη Αβραμόπουλο, θα παρουσιάσουμε σειρά προτάσεων επί κάτι που συζητήσαμε προηγουμένως εδώ και ε, αν συμφωνείτε με τα χαράς να έρθω και να σας εξηγήσω το θέμα από τη στιγμή που θα υποβληθούν οι προτάσεις αύριο όποτε μπορείτε. Δηλαδή ουσιαστικά, πρακτικά αυτό σημαίνει αρχές του επομένου έτους. Ε, ευχαριστώ και συγγνώμη που μακρηγόρησα λίγο. Ευχαριστώ Επίτροπε για αυτή την σύνοψη και ευχαριστούμε που μας υπενθυμίσατε πόσο καλή δουλειά κάνουν τα μέλη της ε, Επιτροπής μας σε διάφορα θέματα. Σήμερα έχουμε μια ψηφοφορία ε, για, το, ε, για την ομοποίηση παρανόμων, παρανόμων εσόδων, για παράδειγμα. Είναι τεράστιο το έργο το οποίο έχει επιτελεστεί. Θα δώσω το λόγο στους αδέλφους. Θα ήθελα να ξεκινήσω εγώ με μια ερώτηση σε ό,τι αφορά την κλίμακα Μπορώ, μου επιτρέπετε, μια γρήγορη ερώτηση. Είδα κάποιους να μορφάζουν. Ε, ε, σε ό,τι αφορά τις ε, συναντήσεις προετοιμασίας, για το πώς εργάζονται τα διάφορα, ε, πώς βλέπουν τα διάφορα μοντέλα για την κλίμακα. Πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή σε ό,τι αφορά το πόσο σημαντικό είναι το πρόβλημα σε ό,τι αφορά το εξτρεμιστικό περιεχόμενο επιγραμμικά. Ε, που, πόσο, σε, σοβαρό είναι το πρόβλημα και πού βρισκόμαστε σε ό,τι αφορά την ε, παρακόλληση διάδοση προπαγάνδας και την ανακατεύθυνση. Ε, ε, είχαμε παρανοήσει το πόσο σημαντικές είναι αυτές οι μέθοδοι ε, για την καταπολέμηση της διάδοσης του τρομοκρατικού αφηγήματος, διότι αυτοί δεν στοχοποιούν εμάς, στοχοποιούν πολύ συγκεκριμένα κοινά, συγκεκριμένο κοινό και ομάδες του πληθυσμού. Αυτή είναι η δική μου ερώτηση. Η κυρία Γκρίσμπεκ ε, είναι πρόεδρος της Υποεπιτροπής Τρομοκρατίας ε, και θα ξεκινήσω από τους συντονιστές, ε, το ΕΛΚ και λοιπά. Γκρίσμπεκ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ναταλία, Ναταλή, συνέχισε. Είπα να ξεκινήσουμε τους συντονιστές τελικά, αλλά ε, όλοι είναι πολύ ευγενικοί ή κουρασμένοι. Ναταλή συνέχισε ως πρόεδρος της Επιτροπής ΤΕΡ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ τον Επίτροπο που είναι παρόν εδώ μια Δευτέρα απόγευμα βράδυ στην, στο ξεκίνημα της Συνόδου. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και για την παρουσία σας λοιπόν, αλλά και για την παρουσία σας γενικά σε όλη την Ευρώπη, αυτό τον τελευταίο καιρό, σε ό,τι αφορά την, ε, ε το πώς χειρίζεστε τα θέματά σας και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Άκουσα πολύ προσεκτικά την παρουσίασή σας, διάβασα και τη σύνοψη της ε, ε συνάντησης ε, του διαλόγου για την ασφάλεια και ήμουν και παρούσα σε ένα τμήμα της ε, συνεδρίασης του Φόρουμ την περασμένη εβδομάδα. Πολλά ενθαρρυντικά μηνύματα βγήκαν από εκεί σε ό,τι αφορά την ικανότητα, τη συλλογική μας ικανότητα να προχωρήσουμε τόσο γρήγορα όσο και αυτοί οι οποίοι διαδίδουν τα συγκεκριμένα μηνύματα της τρομοκρατίας ε, οι οποίοι δρούν ε, σε δίκτυα σε όλο τον πλανήτη. Θα ήθελα να σχολιάσω ένα από αυτά που είπατε, σε ό,τι αφορά ε, την οικοδόμηση ενός αντιλόγου. Ε, είναι κάτι το οποίο θα μας επιτρέψει να ε, καταπολεμήσουμε την προπαγάνδα των ιδιών της τρομοκρατίας. Βλέπουμε στην Ευρώπη ότι ε, δεν ε, οι, οι, οι τρομοκρατικές πράξεις ε, δεν την χάνουν προετοιμασίας ε, εκεί μακριά που γίνονται οι σειράξεις, αλλά πολύ πιο κοντά σε μας. Θέλω λοιπόν να δω την, την ανάλυση της πρακτικής των κρατών μελών. Τα, όλα τα κράτη-μέλη έχουν εφαρμόσει ε, έχουν αναλάβει πρωτοβουλίες ε, τύπου επίσημες εκστρατείες εναντίον του, της ε, τρομοκρατικής ιδεολογίας με αντίλογο και όπως για παράδειγμα στη χώρα μου με την εκστρατεία Stop Jihadism που έδρασε πολύ θετικά τα άλλα κρατημέλη έχουν παρόμοιες εκστρατείες, παρόμοιες πρωτοβουλίες Και επίσης, κάτι που με ενδιαφέρει ιδιαίτερα και εμένα και άλλα μέλη της ε, Ειδική Επιτροπής Τρομοκρατίας, το εξής. Έτσι όπως βλέπετε εσείς συνολικά την κατάσταση, σε αυτές τις εκστρατείες αντιλόγου υπάρχει κάτι ιδιαίτερα αποτελεσματικό, κάποια βέλτιστη πρακτική, κάτι που να έχει ξεχωρίσει σε σχέση με τις υπόλοιπες ε, ε, πρωτοβουλίες. Ευχαριστώ. Thank you very much. Πρόεδρος, ευχαριστούμε Ναταλή. Ε, πολύ καλή ερώτηση. Στην συνάντηση προετοιμασία πράγματι ε, αναδείχθηκε ότι πρόκειται για ένα θέμα το οποίο το αναλαμβάνουν τα κράτη-μέλη και όχι εμείς. Οπότε είναι ενδιαφέρουσα πράγματι η, η παρατήρησή σας. Μόνικα για το ΕΛΚ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Θα ήθελα να σας πω το εξής. Όπως μας εξήγησε ο Βέλγος ειδικό ο κύριος Σαμράνη, οι σαλαφιστές ξεκινάνε από νωρί, από παιδιά 6 ετών, 7, με πολύ λεπτές ε, μεθόδους ε, προσπαθούν να τα προσελκύσουν και σε κάποιες ε, περιπτώσεις βλέπουμε ότι και ο οικογενειακός και ο κοινωνικός κύκλος επιδρούν. Εν τω μεταξύ διαπιστώσαμε στις επισκέψεις μας ότι όλες οι αρχές των χωρών που επισκεφτήκαμε ε, βλέπουμε ότι τώρα επιστρέφουν πολύ περισσότερα γυναικόπαιδα και η αντιμετώπιση τους είναι ε, διαφορετική. Δηλαδή τα παιδιά εν μέρη έχουν ε, ψυχολογικά τραύματα από την Συρία από το να κάνουν ας πούμε μαθήματα το να κάνουν σχολείο σε στρατόπεδο φύγων μέχρι το να έχουν δει δολοφονίες κτλ. Πράγματα λοιπόν τα οποία οδηγούν σε ψυχολογικά τραύματα και πιθανώς σε ριζοσπαστικοποίηση. Υπάρχει κάποια σκέψη για το τι μπορούμε να κάνουμε με τα γυναικόπαιδα τα οποία επιστρέφουν και έχουν αυτά τα ψυχολογικά τραύματα δεύτερο. αναφερθήκατε στο θέμα της χρηματοδότησης της ε, τρομοκρατίας ε, ε, αναφέρθηκε και στο θέμα των Panama Papers. Έχουμε και δικά μας παραθυράκια εδώ πέρα. Βλέπουμε ότι δεν υπάρχουν παραδείγματο χάρη κράτη-μέλη σε αυτόν τον κατάλογο, ενώ ξέρουμε ότι κάποια από αυτά είναι. Και ξέρετε, ε, το τι ακριβώς ε, εννοώ. Βλέπουμε ότι κάποια κράτη-μέλη είναι πολύ επιφυλακτικά για να συνεννοηθούν σε κάποιους ενιαίους ευρωπαϊκούς κανόνες για να κλείσουν τέτοια κανάλια. Εντάξει, βεβαίω αυτό δεν είναι θέμα μόνο χρηματοδότησης τρομοκρατίας, αλλά είναι ένα τεράστιο φάσμα το οποίο καλύπτει και αυτό Απλά απορώ για το ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν φαίνεται να θέλει να δημιουργήσει ένα πρότυπο το οποίο θα αποκλείει τέτοια πράγματα ή τόσο στο βαθμό του δυνατού. Σας ευχαριστώ, Μπίργκιτ, για τους σοσιαλδημοκράτες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε, και είμαι πολύ κουρασμένη, οπότε θα μιλήσω γερμανικά. Ζητώ συγγνώμη. Πρώτα απ' όλα, ο Επίτροπος Κίνγκ ε, ξεκίνησε να μιλάει για πρόληψη και ξεκίνησε με την χρηματοδότηση της νομοκρατίας. Ε, βεβαίως αυτό είναι ένα πρόβλημα ε, περίπλοκο. Οπωσδήποτε υπάρχουν κάποιες δυνατότητες παρέμβασης, αν το οργανώσουμε σωστά, για όλες τις χρηματικές ροές ε, εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βεβαίως είναι δυσκολότερο να κάνουμε κάτι με χρηματικές ροές από τρίτες χώρες προς τρομοκρατικές ομάδες ε, στην Ευρώπη. Ποιες δυνατότητες υπάρχουν εκεί και γνωρίζουμε από ποιες ε, περιοχές υπάρχουν ιδιαίτερες χρηματικές ροές. Και εδώ πέρα βεβαίως θα υπενθυμίσω ότι και κάποιες δυτικές, όπως λέμε, χώρες χρηματοδότησαν όχι δρομοκράτες, αλλά δικτάτορες. Ε, γιατί όταν μιλάμε για την αιτία της τρομοκρατίας πρέπει στο μέλλον να ρίξουμε μια ματιά γιατί υπάρχουν ασταθή κράτη στο Αφγανιστάν, στο Ιράν, στο Ιράκ, στη Συρία και ποια συμμετοχή είχαν οι δυτικές χώρες σε αυτό. Για την πρόληψη, την καταπολέμηση των βασικών αιτιών της τρομοκρατίας ανήκει ε, άρα και η γενική μας ε, αντιμετώπιση των τρίτων χωρών. Είναι μεγάλη υπόθεση. Πρέπει να αναγνωρίσουμε το τι μπορούμε να κάνουμε έτσι ώστε η τεχνολογία η οποία χρησιμοποιείται για να υπάρξει ριζοσπαστικοποίηση θα είναι υποέλεγχο. Και θυμάμαι εδώ πέρα αυτό το οποίο είχε πει η κυρία Χολμάιερ ε, περί του Βέλγου αστυνομικού, αλλά και αμερικανικές υπηρεσίες μας διηγήθηκαν ότι όποιος θέλει να έχει την δυνατότητα θα πρέπει να απευθυνθεί το συντομότερο δυνατόν σε μικρά παιδιά. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να παρέμβει η αστυνομία αλλά και ολόκληρο το κοινωνικό περιβάλλον. Σχολεία, κοινωνική λειτουργία, εκκλησίες κλπ το θέμα τρομοκρατικών εικόνων και ταινιών στο διαδίκτυο είναι οπωσδήποτε και αυτό σημαντικό και το θέμα των αντίθετων μηνυμάτων. Εγώ θεωρώ ότι η χρηματοδότηση τρομοκρατίας είναι τόσο καλή ώστε τα μηνύματα που πρέπει να εκπέμψουμε θα πρέπει να διαμορφωθούν διαφορετικά ανά κράτος μέλος και ανά ομάδα στην οποία απευθύνονται και δεν είναι δυνατόν να υπάρξει ένα ευρωπαϊκό μήνυμα κατά της ε, τρομοκρατίας αλλά θα ήταν χρήσιμο να μας πει ο Επίτροπος ποιες είναι οι εμπειρίες από τα κράτη-μέλη. Ήδη βεβαίως ε, γνωρίζουμε πόσο χρήσιμο είναι να, κατεβαίνει, να κατεβαίνουν ορισμένα περιεχόμενα και οπωσδήποτε υπάρχουν κάποια πράγματα που μπορούν να κατέβουν και θα έπρεπε, αλλά υπάρχουν και κάποιες γκρίζε ζώνες θα έλεγα. Και εδώ πέρα πρέπει να δούμε πώς είναι η συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα για να εμποδίσουμε το να σβηστούν πράγματα που δεν είναι τόσο ξεκάθαρα εγκληματικά ή τρομοκρατικά. Μια τελευταία παρατήρηση, γιατί ακούγεται συνεχώς η φράση πρόληψη και όχι η παρεμπόδιση των χτυπημάτων. Κάτι το οποίο βεβαίω δεν είναι πάντα δυνατόν. Ε, φαίνεται ότι αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημασία, αλλά δεν έχουν εντύπωση ότι ε, το βλέπουν έτσι ε, όλα τα κράτη-μέλη, αν έχει γίνει κάτι σε ένα κράτος μέλος. Δεν ξέρω αν έχετε συγκεκριμένα νούμερα, αλλά βλέποντας και τον αριθμό του προσωπικού, νομίζω ότι ασχολούμαστε πολύ περισσότερο με πράγματα όπως δεδομένα αεροπορικών επιβατών, ε, αιτιάς, ε, διαλειτουργικότητα. Αλλά το θέμα της πρόληψης ε, και της άπορης ζωσφαστικοποίησης έχει μείνει λίγο πίσω, δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Σας ευχαριστώ, Τζοδίθ, για τους Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε τον Επίτροπο για την παρακολούθηση της οδηγίας ε, κατά της ε, ε, ξεπλήματος παρανόμου χρήματος. θα... Το θέμα αυτό εκκρεμεί εδώ και καιρό και θέλω να μοιραστώ μαζί σας το εξής. Πολύ απογοητευσή επικρατεί, αλλά ιδιαίτερος υπό το φως αυτής της συζήτησης να σας πω το εξής. Ε, η Επιτροπή ΤΕΤ την περασμένη Παρασκευή συναντήθηκε με την Europol και ο διευθυντής μιλούσε για, μια, για την ανάγκη μιας ευρωπαϊκής υπηρεσίας οικονομικών πληροφοριών ακριβώς ε, για να εντοπιστούν αυτοί οι οποίοι χρησιμοποιούν ε, παράνομα, παράνομες προσόδους για να χρηματοδοτήσουν την τρομοκρατία. Και το ελάχιστο το οποίο υπήρχε για αυτό το θέμα στο κείμενο εξαφανίστηκε παρόλο που το ζητάει η Europol επειδή δεν το θέλουν τα κράτη-μέλη. Ε, είναι απογοητευτικό αυτό. Δεν το βλέπω εγώ πιθανά αυτό. Ε, τα κράτη-μέλη τουλάχιστον θα μπορούσαν να έχουν κάτι, ένα, μια μικρή συνεισφορά και αργότερα να υπάρχει μια ρήτρα αναθεώρησης για να ενισχυθεί αυτή η παρουσία. Ε, είναι κακή πολιτικό το μήνυμα που στέλνουμε. Αν θέλουμε να καταπολεμήσουμε την τρομοκρατία θα πρέπει να δράσουμε από κοινού και να αντιμετωπίσουμε το θέμα της χρηματοδότησης αυτών των τρομοκρατικών πράξεων. Τώρα, επιστρέφω στο θέμα της ε, ιδεολογίας τρομοκρατίας. Η προετοιμασία, η συνάντηση προετοιμασίας ε, ήταν εξαιρετική. Πάρα πολύ καλοί ομιλητές. Βέβαια, είναι λίγο δύσκολο να γίνει αυτός ο διάλογος δημοσίως. Το τι λειτουργεί και τι δεν λειτουργεί στην ε, καταπολέμηση. Δεν είναι ένα θέμα το οποίο είναι εύκολο να συζητηθεί δημοσίως. Θα ήθελα λοιπόν να σας θέσω ένα πιο γενικό ερώτημα. Ε, το κατέβασμα του τρομοκρατικού περιεχομένου που βρίσκεται επιγραμμικά γίνεται από το Internet Referral Unit ε, που ε, ειδοποιεί ή προειδοποιεί τους παρόχους ότι τέτοιο περιεχόμενο δεν συνάδει με τις αρχές τους. Την περασμένη Παρασκευή έγινε και μια παρανόηση. Μιλούσαμε με τον Ολλανδό συντονιστή για θέμα τρομοκρατίας η χώρα μου κατεβάζει περιεχόμενο μόνο όταν πραγματικά είναι ε, εγκληματικό, όταν δηλαδή προβλέπεται ποινή. Όμως η ευρωπαϊκή πολιτική είναι λίγο διαφορετική από ό,τι φαίνεται. Μπορείτε να μας το ξεκαθαρίσετε, διότι θα αρχίζα να ανησυχώ αν κατεβάζαμε περιεχόμενο μέσω της ε, αντίστοιχης μονάδας της Europol χωρίς το περιεχόμενο αυτό να είναι εγκληματικής φύσεως. Δηλαδή, αν κάποιος κατέφυγε στο δικαστήριο δεν θα, θα, θα ποινή για αυτό το περιεχόμενο. Τελευταία μου ερώτηση. Η συζήτηση γίνεται ε, πολύ συχνά για το, το αφήγημα της τρομοκρατίας που οδηγεί σε ριζοσπαστικοποίηση. Όμως βλέπουμε σε πολλές χώρες ε, αύξηση και των τρομοκρατικών δράσεων και πράξεων ακροδεξιών οργανώσεων. Τι ακριβώς, γιατί ακριβώς μιλάμε για ποιο ακριβώ αφήγημα μιλάμε, γιατί η ακροδεξιά επίση προβαίνει σε τρομοκρατικέ ενέργειε. Ευχαριστώ. Ο κ. Τζεντόφσκι, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν ήταν σειρά πάρω το λόγο. Βλέπετε, εγώ δεν είμαι κάποιος πρόεδρος επιτροπής, δεν είμαι συντονιστής. Περίμενα υπομονετικά όμως για τη συζήτηση. Χαίρομαι που παρίσταμε. Δυστυχώς δεν μπόρεσα να συμμετάσχω σε αυτή την αποστολή που συζητούμε. Ήμουν στο Νεπάλ, αλλά για τη χρηματοδότηση. Κύριε Επίτροπε, όταν αναφερθήκατε στη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας μέσω bitcoin, από ό,τι κατάλαβα απαντήσατε ότι είναι κάπως Ανόητο αυτό σαν σκέψη. Αυτό ήταν εν είδη απαντήσεω σε ένα ερώτημα δικό μου και συναδέλφου. Όταν κάναμε την ερώτηση αν μπορούν οι τρομοκράτε να χρηματοδοτούνται από εικονικά νομίσματα, διαδικτυακά νομίσματα. Νομίζω ότι θα πρέπει να το σκεφτούμε αυτό από πλευράς νομικής περισσότερο. Μίλησα με εμπειρογνώμονες οι οποίοι ανέφεραν ότι υπήρχε κατασχέθηκε μεγάλο ποσό bitcoin στη Βουλγαρία. Και φαίνεται ότι η Βουλγαρία είναι πολύ πλούσια χώρα σε bitcoin. Θα ήθελα να ξέρω κατά πόσο αυτό το θέμα συζητείτε, προκύπτει, πώς το προσεγγίζετε και πώς θέλετε να αποφύγετε την χρήση του bitcoin ή άλλων εικονικών νομισμάτων, ώστε να μας απειλήσουν. Μπορώ να δημιουργήσω μια εταιρεία στο Ηνωμένο Βασίλειο τάχιστα αυτή είναι η πρώτη μου ερώτηση. Έτσι. Φτιάχνω μια εταιρεία στον Ηνωμένο Βασίλειο. Και μπορώ να βάλω χρήματα σε αυτή την επιχείρηση και μπορώ να χρηματοδοτήσω ό,τι θέλω μέσω τη εταιρεία. Και μετά μπορώ να πω στην Κύπρο και μπορώ να ιδρύσω μια άλλη εταιρεία εκεί. Δεν υπάρχει διαφάνεια. Δεν υπάρχει ανοιχτή διαφανής προσέγγιση για τη λειτουργία των δομών αυτών. Είσαστε έτοιμος να καταπολεμήσετε αυτά τα φαινόμενα και αν ναι, πώς. Τι είναι η τρόπο. Η χρηματοδότηση τρομοκρατίας την αναφέρατε. Έχω μια συγκεκριμένη ερώτηση. Πρόσφατα είχαμε την επέτειο της επιθέσεως κατά το Τσάλι Εμπντό, της τρομοκρατικής επιθέσεως. Και είδαμε ότι τα αδέλφια που διέπραξαν την επίθεση είχαν ριζοσπαστικοποιηθεί, τουλάχιστον ένας από αυτούς είχε ριζοσπαστικοποιηθεί, ενώ ήταν στη φυλακή. Λοιπόν, ήταν επίσης στον κατάλογο ε, εκείνων που δεν επιτρέπεται να ταξιδέψουν αεροπορικός Οι γαλλικές μυστικές υπηρεσίες όμως δεν τον παρακολούθησαν και είπαν ότι δεν είχαν αρκετά χρήματα για να παρακολουθούν τους πάντες. Αυτή ήταν η απάντησή τους. Και τελικά αυτός ο τρομοκράτης δεν έκανε τίποτα προφανές για να ε, προσελκύσει τις ε, υποψίες, να δημιουργήσει υποψίες. Όμως πραγματοποίησε την επίθεση. Πώς το βλέπετε αυτό. Έχουμε λίστες αλλά μετά δεν έχουμε αρκετού πόρου για να παρακολουθούμε όλου αυτού οι οποίοι βρίσκονται στις λίστες. Τελευταία ερώτηση. Υποτεθείστε ότι είσαστε από μια μικρή χώρα της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και... Έχετε 3.000 αναφορές στο, στο λογαριασμό σας Facebook ε, με απειλές. Θα σε κρεμάσουμε, θα κρεμάσουμε εσένα και όλη την οικογένειά σου, όλους αγαπητούς. 3.000 χτυπήματα. Και α πούμε ότι είσαστε ένα ευρωβουλευτή που το αναφέρατε αυτό. Και εντό μια εβδομάδα δεν παίρνετε καμία απάντηση, τίποτα. Και παρόλο που υπάρχουν εικόνες που παρουσιάζονται ανθρώπων στην κρεμάλα, η απάντηση είναι ότι δεν, δεν τρέχει τίποτα. Σε τέτοιε περιπτώσεις πιστεύετε ότι θα μας εμπιστεύεται ο κόσμος, θα πιστέψει ότι πραγματικά προσπαθούμε να καταπολεμήσουμε την τρομοκρατία, θα πιστεύετε θα γελούν τελικά αυτοί που χρησιμοποιούν το Facebook. Μάλλον αυτοί που έχουν το Facebook τελικά δεν μας πούν στα σοβαρά. Μάλλον μα κοροϊδεύουν. Αυτό είναι το συμπέρασμα. Τι πιστεύετε εσεί. Να πω ότι στην προπαρασκευαστική συνεδρίαση είχαμε καλέσει την Google, αλλά τελευταία στιγμή είχαν ένα κόλλημα. Τώρα αναφέρω αυτό για τη συμμετοχή του κλάδου. Κυρία Μαϊτέ ε, Θέλω να ευχαριστήσω τον Επίτροπο καταρχήν για την έκθεση που μας παρουσίασε, ε, τη σύνοψη αυτή που έκανε, ε, την δομημένη του παρουσίαση. Η μια συνάδελφος μίλησε πριν από μένα, είπε και νομίζω ότι έχει δίκιο, ότι το επιχειρηματικό κομμάτι αναπτύσσεται πολύ πιο επαγγελματικά και γρήγορα από ότι το κομμάτι της πρόληψης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει περισσότερους ε, πόρους ε, και γι' αυτό το λόγο ε, λειτουργεί καλύτερα το επιχειρησιακό κομμάτι, αλλά τα κράτη-μέλη χρειάζεται να κάνουν περισσότερες προσπάθειες για την πρόληψη. Βέβαια, έχουν ξεκινήσει αρκετέ ε, ε, πρωτοβουλίε τον τελευταίο καιρό, δεν έχουμε όμω μια πλήρη κάλυψη. Ε, το, η μέθοδος της ανακατεύθυνσης, η, ε, συνεργασία με τον Google και άλλους παρόχους κλπ. Ε, νομίζω ότι... Α, 7 Δεκεμβρίου έχουμε και το πρώτο tweet, κάτι πολύ καινούριο. Και επί τη να πω ότι κανένα δεν ξέρει ακριβώ ποιο είναι πίσω από αυτά τα tweet και αυτό μπορεί να δημιουργήσει ανασφάλεια. Μετά, μιλήσατε για, τα... για του πόρου που χρησιμοποιούν τα τελευταία χρόνια, καινούρια πράγματα προκύπτουν. όλα αυτά τα χρήματα, όλο αυτό το σχετικά άτυπο σύστημα πρόληψης. Θα ήθελα να ξέρω, θα, θα γίνει, θα αξιολογηθεί ως προς την αποτελεσματικότητά του στο μέλλον για το πόσο πραγματικά προλαμβάνει ε, αυτές τις τρομοκρατικές πράξεις. Η κατάρτιση των εκπαιδευτών επίσης είναι πολύ σημαντικό να γίνεται σωστό, σωστά. Ε, δεν θέλουμε απλώς ανθρώπους που έχουν ε, πάθος ε, χωρίς γνώσεις, έτσι, επειδή μόνο ε, θέλουν να πολεμήσουν αυτούς τους ακραίους τρομοκράτες κλπ. Όχι, θέλουμε ανθρώπους πραγματικά να έχουν κατάλληλα προσόντα. Παρακαλώ συνεχίστε προκειμένου να διαρθρωθεί καλύτερα η δράση μας για την πρόληψη και προκειμένου με εξίσου δομημένο τρόπο να αντιμετωπίζουμε τις διάφορες πραγματικότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι μόνο μερικές. Οι εκπαιδευτές ιδιαίτερως θα πρέπει να είναι άτομα που να έχουν εμπειρία, πρακτική εμπειρία. Ευχαριστώ. Mr. Ευχαριστώ Ντιούρεκ. Ε, ε, ε, ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Επίτροπε για τις πληροφορίες που μας δώσατε. Είπατε ότι πρέπει να εστιάσουμε στις ομάδες εκείνες που είναι πιο ευεπίφορες στην ριζοσπαστικοποίηση και πρέπει να ασχοληθούμε με τις αιτίε. Έχουμε και εμείς κάποιες σχετικές απόψεις. Προσπαθούμε να ενημερώσουμε τις πληροφορίες μας. Το θέμα είναι πώς θα βρούμε και θα ταυτοποιήσουμε αυτές τις ε, ομάδες για να προλάβουμε επίσης ε, και τις αιτίες ε, της τρομοκρατία, όπως λέτε. Σας ευχαριστώ. Βεβαίω είναι πάρα πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστεί το αφήγημα όταν τα κράτη-μέλη δεν κάνουν τίποτα για να προωθήσουν την ένταξη. Μέσω κοινωνικής ε, ένταξης και τα λοιπά. Αλλά το ερώτημά μου είναι το εξής. Σε ποιο βαθμό ένα αφήγημα δεν βοηθείται από το ότι τα κράτη-μέλη μας επιτρέπουν σε χώρες όπως η Αραβία και άλλες να πληρώνουν για τους ημάμιδες ε, στα τζαμιά και αλλού και σε ιεροδιδασκαλία με ντρεσέδες και τα λοιπά. Μιλάμε για μια διάδοση των πιο ακραίων ε, απόψεων που ανοίγουν τον δρόμο για την ριζοσπαστικοποίηση. Και μια που αναφέρατε την χρηματοδότηση της ε, τρομοκρατίας. Η ομάδα μας ε, την προηγούμενη εβδομάδα πήγε στην Χάγη και συνάντησε την Europol. Το είπε η Ιουδίθ και εσείς ότι το θέμα μιας ευρωπαϊκής μονάδας ε, πληροφο... οικονομικών πληροφοριών ε, έχει μεγάλη σημασία. Δεν έχει νόημα να περάσουμε σε άλλη μια οδηγία αν δεν ε, έχουμε κάτι το ουσιαστικό. Μια Ευρωπαϊκή Μονάδα Οικονομικών Πληροφοριών το θέμα της διαφάνειας ε, για τα καταπιστεύματα και θα έλεγα το θέμα της ταυτοποίησης των οχημάτων ειδικού σκοπού που έρχονται και δραστηριοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά δεν το θέλουν αυτό τα κράτη-μέλη. Το είπε και η Τζούντιθ και λέει ότι είναι θέμα κυριαρχίας. Μα όχι, δεν είναι θέμα κυριαρχίας. Είναι θέμα προστασίας των διεφθαρμένων, των εγκληματιών και μεταξύ αυτών των τρομοκρατών. Εάν επιτρέψουμε λοιπόν αυτό το αφήγημα της κυριαρχίας των κρατών μελών θα έχουμε μια πέμπτη οδηγία η οποία πραγματικά θα αξίζει το χαρτί στο οποίο θα έχει τυπωθεί. Και αυτό το μήνυμα πρέπει να ακουστεί κάθαρα από την Κομισιόν και από εμά όμως, εμάς που καθόμαστε στην σχετική διαπραγματευτική ομάδα και να ακουστεί καθαρά στα κράτη-μέλη. Είναι θέμα καταπολέμησης της τρομοκρατίας, του οργανωμένου εγκλήματος που στηρίζει την τρομοκρατία τέλος θα ήθελα να σας ρωτήσω τι κάνει η Κομισιόν για να εξετάσει τον ρόλο των κρυπτονομισμάτων και όχι μόνο του bitcoin και μάλιστα ε, ε, για την διευκόλυνση της χρηματοδότησης του οργανωμένου κλίματος και της τρομοκρατίας και θα ήθελα να ρωτήσω αν έχει υπάρξει κάποια συνεννόηση με τον Επίτροπο Μοσκοβισή που έχει μια πάρα πολύ σημαντική έκθεση για το πώς χρησιμοποιείται ο ΦΠΑ για τη χρηματοδότηση τρομοκρατικών δραστηριοτήτων ακόμα και από την Αλκάιντα. Σας ευχαριστώ. Um, κυρία Βερζιά. Υπάρχει κάποιος άλλος μετά την κυρία Βερζιά. Μου να ξέχασα τελευταία που το λόγο κυρία Βερζιά. Ευχαριστώ. Ζητώ συγγνώμη κύριε Επίτροπε, διότι έχασα σχεδόν όλη σας την παρέμβαση. Βλέπετε όμως έπρεπε να είμαι σε άλλη συνεδρίαση. Θέλω να πω καταρχάς ότι όσο προχωρούμε στο έργο που κάνουμε για το θέμα, εδώ, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή αλλού, και στις διάφορες συναντήσει που έχουμε τόσο γνωρίζουμε ότι δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις, ότι υπάρχουν διαφορετικές οπτικές γωνίες και ετερογένειες όσον αφάτη την προσέγγιση. Ακούγοντας τα κράτη-μέλη, έχουμε την εντύπωση ότι αισθάνονται ότι παρεμβαίνουμε στην εθνική τους κυριαρχία με αυτά τα μέτρα. Ταυτόχρονα, παραλλήλως, υπονομεύεται και η θέση της Ευρωπαϊκής Ενώσης σε αυτό το θέμα. Είναι πολύ εύκολο να κατηγορείται η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία δεν κάνει το καθήκον της. Όλα αυτά μας βοηθούν να έχουμε ένα πολύ συνοπτικό αφήγημα και περιοριστικό και υπεραπλουστευμένο και αυτή η απλούστευση μιλήσαμε αποφυγή της ρίζοσπαστικοποίησης κλπ. Αλλά αυτή η περαπλούστευση είναι ασύμβατη με την ισορροπία. Ισορροπία μεταξύ της ανάγκης για ασφάλεια και της ελευθερίας. Όποια και είναι αυτή. Ανησυχώ ακόμα περισσότερο ακούγοντας κάποιους συναδέλφους που πιστεύουν ότι είχαμε αποφύγει τα χτυπήματα στη Γαλλία, αν είχαν περισσότερα χρήματα οι Γάλλοι αστυνομικοί και μυστικές υπηρεσίες να παρακολουθούν καλύτερα τους υπόπτους. Μιλήστε μας λίγο για την ισορροπία μεταξύ ασφαλείας και ελευθερίας. Ασφαλείας για την καταπολέμηση τρομοκρατίας και ελευθερίας μεταξύ των δύο. Είμαι Γαλλίδα, έχω κάποιες ανησυχίες για το θέμα μετά τον πρόσφατο νόμο ψηφίστηκε στη χώρα μου. Μετά πάνω στο ερώτημα της Άννα για τη συνεργασία με τρίτες χώρες. Αναφέρθηκε στις χώρες του κόλπου. Ανησυχώ και μάλιστα μετά την αποστολή που κάναμε στη Γαλλία, ανησυχώ για τη συνεργασία με την Τουρκία. Διότι όλοι γνωρίζουμε ότι ο ορισμός της τρομοκρατίας από πλευράς Τουρκίας είναι τουλάχιστον δύσκολος, περίπλοκος. Και πολλά άτομα αυτή τη στιγμή που είναι στις φυλακές της τουρκικές στα πλαίσια καταπληκτικής τρομοκρατίας δεν έχουν καμία σχέση αυτοί οι άνθρωποι με την τρομοκρατία. Και κατά κάποιο τρόπο αυτό με οδηγεί στο προηγούμενο ερώτημα. Όταν συνεργαζόμαστε με τίτες χώρες, πρέπει να προσέχουμε τι γίνεται με το θέμα της ελευθερίας. Και μάλιστα με χώρες οι οποίες δεν προστατεύουν επαρκώς την ελευθερία. Ευχαριστώ. Αυτό ήταν ο τελευταίος. Κάποιος άλλος θέλει να πάρει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Το λόγο. Ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις σας και για την ε, προσήλωσή σας στο έργο σας. Θα προσπαθήσω να απαντήσω όσο μπορώ. Αν ε, δεν πάρετε απάντηση, ελάτε να με δείτε. Ή επικοινωνήστε μαζί μου. Εσείς πρόεδρε ξεκινήσατε με μια γενική ερώτηση για το μέγεθος του προβλήματος ε, στο διαδίκτυο. Δεν θα αποφύγω την απάντηση. Νομίζω ότι τα καταφέρνουμε καλά και σε ό,τι αφορά το κατέβασμα περιεχομένου. Ε, εκεί έχουμε δεκάδες χιλιάδες περιπτώσεις και καλά με τις ε, εταιρείε, τους ε, ε, παρόχους που βελτιώνουν τα δικά τους εργαλεία εντοπισμού τέτοιου περιεχομένου. Όμως, ξεκολουθούμε να έχουμε εκατοντάδες χιλιάδες ακόμα ε, περιπτώσεις περιεχομένου που βρίσκονται στο διαδίκτυο ακόμα. Οπότε είναι μεγάλη η πρόκληση τόσο ό,τι αφορά το μέγεθος όσο και τόσο ό,τι αφορά την ταχύτητα. Δηλαδή τον όγκο και την ταχύτητα. Σε ό,τι αφορά την ταχύτητα. Όσο, όσο κάτι παραμένει στο διαδίκτυο, τόσο πολύ μπορεί να διαδοθεί και να αυξηθεί η, το, ε, η επίδρασή του. Το σημαντικό είναι αυτό που λέμε η πρώτη ώρα. Πρέπει να κατεβαίνει αυτό το περιεχόμενο το συντομότερο δυνατόν. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον όγκο, όση πρόοδο και να κάνουμε με τις μεγάλες πλατφόρμες, υπάρχει ένα θέμα μετανάστευσης σε άλλες μικρότερες πλατφόρμες. Η Ευρωπόλ εργάζεται σε 100 πλατφόρμες αυτή τη στιγμή περίπου, εντόπισε περιεχόμενο σε 150 πλατφόρμες. Δεν θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το, τα θέματα όλων σε όλες τις πλατφόρμες. Υπάρχουν πλατφόρμες που συνδέονται πάρα πολύ με το Ισλαμικό κράτος ε, που τις έχουν δημιουργήσει και τις διαχειρίζονται οι άνθρωποι που δημιουργούν το περιεχόμενο. Είναι πολύ δύσκολο να εισέλθουμε σε αυτές τις πλατφόρμες. Όμως, σίγουρα μπορούμε να βελτιώσουμε το αποτέλεσμά μας συνεργαζόμενοι και στηρίζοντας το οικοσύστημα άλλων πλατφορμών. Μπορούμε να βελτιώσουμε τη δράση μας από τη στιγμή που εντοπίζεται το περιεχόμενο ε, έτσι ώστε οι διοκτικές αρχές να μπορέσουν να δράσουν γρήγορα. Επίσης θα πρέπει να βελτιωθούμε στην παρακολούθηση του τι κάνουμε, στη μέτρηση των αποτελεσμάτων, διότι ε, το όλα βασίζονται στο feedback που παίρνουμε από τους συνεργάτες μας. Η Europol κάνει πολύ καλή δουλειά, ορισμένα κρατημέλη κάνουν επίσης πολύ καλή δουλειά, έχουν ολόκληρη, ε, ολόκληρες δομές εντοπισμού ε, περιεχομένου και ε, οι συνεργάτες μας στις πλατφόρμες. Όλα αυτά θα πρέπει να τα βάλουμε στην ίδια εικόνα έτσι ώστε πραγματικά να δούμε ποιο είναι το πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή το μέγεθος είναι αρκετά μεγάλο. Σωστά θέσατε το ερώτημα. Υπάρχει κάτι άλλο στο οποίο θέλω να επιστρέψω και το σχολίασαν και άλλοι. Κυρία Σαρτζεντίνη για παράδειγμα. Σε τι εστιαζόμαστε. Σε πρώτη προσέγγιση, και αυτό είναι σαφές από το έργο της Europol αλλά και των εθνικών ε, μονάδων εστιάζονται σε παράνομο περιεχόμενο ή περιεχόμενο το οποίο ενθαρρύνει παράνομες δράσεις και πράξεις. Σε ό,τι αφορά την τρομοκρατία, έχουμε συμφωνήσει για το τι είναι παράνομο. Για παράδειγμα, εκπαίδευση, στρατολόγηση, ενθάρρυνση ατόμων να ταξιδέψουν σε ζώνες σειράξεων είναι πράγματα τα οποία θεωρούμε ότι θα πρέπει να κατεβαίνουν από το ίντερνετ. Όπως και οτιδήποτε βέβαια προτρέπει σε τρομοκρατικές πράξεις. Όλα αυτά πρέπει να τα αναλαμβάνουν οι μονάδες αναφοράς διαδικτυακού περιεχομένου. Οπότε σε αυτά εστιάζουμε καταρχήν. Γιατί Αυτά ε, είναι μέτρα τα οποία έχουμε συμφωνήσει. Ορισμένες χώρες έχουν και τη δική τους εθνική νομοθεσία επιπλέον, κάτι το οποίο δεν είναι εναρμονισμένο. Η ευρωπαϊκή νομοθεσία, ναι, έχει εναρμονιστεί σε όλα τα κράτη-μέλη. Αυτός ο κοινός παρανομαστής. Σε δεύτερο επίπεδο, αφού εντοπιστεί το περιεχόμενο, είναι αλήθεια, απαντώντας στην κυρία Σαρτζεντίνη, ότι η Europol όταν αναφέρει το περιεχόμενο αυτό στις πλατφόρμες το συζητά μαζί τους για να μάθει ποια είναι η άποψη της ίδιας της πλατφόρμας για αυτό το περιεχόμενο ε, συμμορφώνεται με τους κανόνες της. Αυτή, αυτό είναι κάτι που γίνεται σε συνεργασία με τις πλατφόρμες. Διότι και αυτοί έχουν τους δικούς τους κανόνες και εμείς έχουμε τους, τα δικά μας κριτήρια για, τις, για την αναφορά διαδικτυακού περιεχομένου. Οπότε πρέπει να δούμε αν αυτά συνάδουν. Φαντάζομαι ότι γι' αυτό σας μίλησε η Europol και αυτό είναι πολύ σημαντικό για να χτίσουμε μια σχέση συνεργασίας με τις πλατφόρμες. 80-90% του περιεχομένου που αναφέρεται από την Europol από τις εθνικές μονάδες κατεβαίνει τελικά από το ίντερνετ. Και δεν μιλάμε για περιεχόμενο το οποίο το έχει δημιουργήσει κάποια ε, ακραία μουσουλμανική οργάνωση. Ε, μιλούμε και για περιεχόμενο ακροδεξιών οργανώσεων. Ε, στην πράξη βέβαια το μεγαλύτερο όγκος περιεχομένου είναι ε, Ισλαμικής προέλευσης. Ισλαμιστικής προέλευσης να το πω έτσι. Ε, δεν είναι όμως ότι εστιάζουμε σε αυτό. Ε, έχουμε περισσότερο τέτοιο περιεχόμενο που κατεβαίνει επειδή ακριβώς είναι μεγαλύτερος όγκος τέτοιου περιεχομένου που υπάρχει στο διαδίκτυο. Τώρα, σε ό,τι αφορά την αποτελεσματικότητα του αντιλόγου μας, το ρώτησε η κυρία Κρίσπεκ, είναι μεγάλη ε, πρόκληση αυτή στην αξιολόγηση της ε, πρόληψης κάθε φορά, όλες, σε όλες τις περιπτώσεις, είναι δύσκολο να δούμε πόσα, πόσο ακριβώς επιτυχημένοι ήμασταν. Συμφωνώ με τον συνάδελφο δίπλα σας που είπε πως η πρόκληση είναι, η, το πρόβλημα είναι να συνδέσουμε την αξιολόγηση με την πραγματική εμπειρία. Στην Βόρεια Ιρλανδία για πολλά χρόνια προσπαθήσαμε να αποφύγουμε την ζωσπαστικοποίηση με πρόληψη. Άλλο το περιβάλλον, αλλά ορισμένες από τις τεχνικές είναι ίδιες. Για παράδειγμα, ε, πολλοί νέοι υφίσταντο, να το πούμε έτσι, ε, μια ιδεολογική ε, πίεση από μεγαλύτερους να κινηθούν προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Δεν μπορώ να σας πω ποια ήταν η επιτυχία, αλλά μπορώ να σας πω ότι οπωσδήποτε πρέπει να γίνουν τέτοια προγράμματα. Ανεξαρτήτως του αν τελικά θα καταφέρουμε να πείσουμε ή να αποτρέψουμε έναν ή δύο μόνο. Αν αυτό πρέπει να γίνει βέβαια στο ίντερνετ και όχι στις φυλακές, στα σχολεία, γίνεται ακόμα πιο δύσκολο να μετρήσουμε την αποτελεσματικότητα. Πρέπει λιγάκι να δούμε το θέμα εμπειρικά. Οπότε η κυρία Κρίσπεκ ρώτησε, έχουν ξεκινήσει κάτι παρόμοιο όλα τα κράτη-μέλη. Δεν είμαι σίγουρος ότι όλα τα κράτη-μέλη έχουν ξεκινήσει. Ορισμένα κράτη-μέλη αντιμετωπίζουν πιο σοβαρά προβλήματα από ό,τι άλλες. Αυτά τα κρατημέλη τα οποία έχουν εμπειρία και καταλαβαίνουν το μεγάλο, τον, το, την κλίμακα του προβλήματος έχουν κάνει πολλή δουλειά. Για παράδειγμα το Stop Jihad πράγματι είναι ένα πρόγραμμα το οποίο ήταν πολύ καλό και είναι παράδειγμα. Και στο Βέλγιο υπάρχουν προγράμματα. Υπάρχει και ένα γερμανικό πρόγραμμα, το Life Democracy, σε ομοσπενδιακό επίπεδο, αν έχω καταλάβει καλά, προσαρμοσμένο στι συνθήκε τη Γερμανίας. Στη Βρετανία υπάρχουν πολλά μοντέλα, ορισμένα μπορεί να είναι χρήσιμα αλλού, αλλά όχι όλα απαραίτητα. Έχουν σχεδιαστεί για συγκεκριμένε καταστάσεις και συνθήκες. Στις κάτω χώρες υπάρχει η πρωτοβουλία Speak Up, που απευθύνεται σε νέους κυρίως. Πολύ καλή και αυτή. Δεν νομίζω όμω ότι υπάρχει ένα μοντέλο το οποίο να κάνει για όλου και για όλε τις περιστάσει. Ακόμα και όταν μιλάμε και για, μόνο για το ίντερνετ, πάλι θα πρέπει ε, να σχεδιάσουμε πράγματα τα οποία να μπορούν να προσαρμοστούν, να είναι προσαρμοσμένα σε διαφορετικέ καταστάσει. Σίγουρα πιστεύω πως πρέπει να συνεργαστείτε με, τις, ε, με τον κλάδο. Είπατε ότι προσκαλέσατε την Google και δεν κατάφεραν να έρθουν. Θα πρέπει να τους ξαναπροσκαλέσετε. Είναι πολύ σημαντικό γιατί αυτοί πραγματικά εργάζονται πάρα πολύ καινοτόμα για το πώς μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις τεχνικές τους και την γνώμη τους, τη γνώση τους για να ανακατευθύνουν άτομα τα οποία αναζητούν τέτοιο περιεχόμενο ακραίο. Ναι, ήταν να έρθουν και ε, το ακύρωσαν τελευταία στιγμή κάτι του συνέβη. Δεν νομίζω ότι είχαν κακή πρόθεση. Όχι, ούτε εγώ το είπα αυτό. Δεν τους επέκρινα. Νομίζω ότι κάνουν πολύ καλή δουλειά στην Google προκειμένου άτομα τα οποία αναζητούν τέτοιου είδους υλικό που τους οδηγεί σε ζωοσπαστικοποίηση να τους ανακατευθύνουν σε άλλο υλικό το οποίο έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να θέτει κρίσιμα ερωτήματα σε αυτούς τους ανθρώπους. Τέτοιου είδους πρωτοβουλίες νομίζω ότι πρέπει να αποτελέσουν τη μαγιά για τη δουλειά των υπολείπων. Κάποιοι αναφέρθηκαν στις δραστηριότητες τρίτων χωρών, σαλαφιστικές δραστηριότητες, χρηματοδότηση από τρίτες χώρες κλπ. Γνωρίζουμε ότι η χρηματοδότηση από τρίτες χώρες πραγματικά ε, επηρεάζει την κατάσταση και έχουμε συζητήσει στην Κομισιόν με ανθρώπους που εργάζονται σε τέτοια θέματα. Σας λέω ένα παράδειγμα. Ε, πήγαμε στο Μόλεμπεκ, ε, στην Βελική πρωτεύουσα και είδαμε τους ανθρώπους που στην πράξη ασχολούνται με τέτοιου θέματα. Είναι δύσκολο όμως να δούμε τι μπορεί να γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να αντιμετωπιστούν τέτοια θέματα τα οποία έχουν άμεση σχέση με κρατικές αρχές που σχετίζονται με θρησκευτικέ αρχέ που είναι και πάλι διαφορετικέ από χώρα σε χώρα. Δεν μπορούμε να το αγνοήσουμε κιόλα. Ούτε και αγνοούμε την πρόκληση που αντιπροσωπεύουν οι, οι επιστρέφοντες από ταξίδια σε ε, χώρες ε, που, που επικρατούν σειράξεις και μπορεί να ε, διασπείρουν μηνύματα ρίζοσπαστικοποίησης ακόμα και αν οι ίδιοι δεν εμπλακούν σε τρομοκρατικές πράξεις. Πέρσι το καλοκαίρι δημοσιεύτηκε μια μελέτη για όλες ε, τις πτυχές αυτών των προβλημάτων ε, γιατί τα προβλήματα των επιστρεφόντων δεν είναι μόνο αστυνομικά είναι θέματα ένταξης είναι θέματα ε, εκπαίδευσης, είναι κοινωνικά θέματα, ε, είναι θέματα τα οποία μπορεί να προκύψουν από την διάδοση υλικού που οδηγεί σε ριζοφυστικοποίηση κλπ. Οπότε είναι σημαντικό να εστιάζουμε και σε αυτά τα ζητήματα. Και δεν είναι μόνο οι νέοι οι ευάλωτες ομάδες. Με ρωτήσατε πώς μπορούμε να εντοπίσουμε τις ευάλωτες ομάδες. Δεν είναι μόνο οι νέοι. οι, οι ειδικοί έχουν πολύ συγκεκριμένη εμπειρία, ξέρουν ότι σίγουρα είναι πολλοί νέοι, αλλά όχι μόνο οι νέοι, δεν είναι μόνο νέοι. Είναι άτομα που βρίσκονται σε φυλακέ, άτομα που είναι εκτό του εκπαιδευτικού συστήματο, πρώην φυλακισμένοι, συγκεκριμένε ομάδε, οι οποίε όμω δεν είναι οι μοναδικέ. Γι' αυτό το λόγο το δίκτυό μα έχει δομηθεί με τρόπο που επιτρέπει στους ε, ειδικού που εργάζονται στο πεδίο ε, να ανταλλάσσουν πρακτικές και γνώση. Η ενσωμάτωση είναι ένα τμήμα της ε, πρόκλησης που έχουμε κυρία Γκόμες και στην Κομισιόν σήμερα, λίγο νωρίτερα σήμερα, συζητήσαμε ακριβώς το πώς μπορούμε οριζόντια στην Κομισιόν να συντονίσουμε τα κονδύλια της εκπαίδευσης, της, ε, ε, του πολιτισμού ε, και τα κοινωνικά κονδύλια εργασιακά, ε, απασχόλησης κλπ. έτσι ώστε να καταπολεμήσουμε ταυτόχρονα με τα ίδια κονδύλια και τη ριζοσπαστικοποίηση. Να πω κάτι άλλο για τις τρίτες χώρες. Υπάρχει μία πρόκληση για τις τρίτες χώρες από άτομα που τρέφουν. Η διάλυση του λεγόμενου Ισλαμικού κράτους ε, επιτόπου έχει ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση για ανθρώπους οι οποίοι ίσως θέλουν να επιστρέψουν στην Ευρώπη και δικαίως με έχετε ξαναρωτήσει για αυτό στο παρελθόν αλλά αρκετοί από τους ε, μαχητές ε, που βρέθηκαν σε Ιράκ και Συρία δεν ξεκίνησαν από την Ευρώπη, ξεκίνησαν από άλλες χώρες και υπάρχει το ζήτημα επιστροφής ε, των ανθρώπων αυτών σε αυτές τις χώρες ή του να πάνε αλλού σε άλλα μέρη όπου υπάρχει αστάθεια είτε μιλάμε για Αφγανιστάν, η Εμένη ή η Λιβύη έχουμε νομίζω εμείς συμφέρον να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε χώρες ειδικά στη γειτονιά μας που επηρεάζονται από προβλήματα από ανθρώπους που επιστρέφουν από το Ιράκ και την ε, Συρία. Γι' αυτό ακριβώς προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα δίκτυο διαλόγου πόλεων, γι' αυτό έχουμε προγράμματα που εστιάζουν στην ενίσχυση της ασφάλειας, στην καταπολέμηση της ε, τρομοκρατίας, ε, ειδικά στην γειτονιά μας και θεωρούμε ότι γύρω στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ εξωτερικών προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν μια διάσταση ασφάλειας που έχει μεγάλη σημασία για αυτήν την ε, δουλειά. Κάνοντας αυτά τα πράγματα, για να απαντήσω δηλαδή και στο ερώτημα της κυρίας Βερζιά, ε, με την Τουρκία ή με οποιαδήποτε άλλη χώρα, φροντίζουμε βεβαίως πάντα η συνεργασία μας να βασίζεται στις αρχές μας. Δεν θα προωθήσουμε μια συνεργασία η οποία υπονομεύει τις αρχές μας να... Α, ναι, να πάω λίγο στο bitcoin πριν περάσω στο ευρύτερο ζήτημα του ξεπλήματος χρήματος. Για το συγκεκριμένο θέμα το οποίο μας ρωτήσατε για το bitcoin ως ε, χρηματοδότη της ε, τρομοκρατίας το γνωρίζουμε. Ε, πρώτα απ' όλα, αν γίνει κάτι με το bitcoin παράνομο, πρέπει να το αντιμετωπίσουμε ούτως ή άλλως. Αλλά ειδικά εστιάζουμε στο bitcoin και στα άλλα εικονικά νομίσματα ως ε, έναν τρόπο διευκόλυνσης ε, της ε, εγκληματικότητας και πιθανώς της τρομοκρατίας. Γι' αυτό ακριβώς έχουμε κάνει μια σειρά συνεδρίων για το πώς θα ενισχύσουμε την καταπολέμηση της ε, κατάχρησης των νομισμάτων αυτών για ξέπλυμα χρήματος, ε, τρομοκρατία κτλ. Και οπωσδήποτε μπορώ να σας στείλω και τις σχετικές, ε, τα συμπεράσματα των σχετικών συνεδρίων. Για τα ερωτήματα τώρα τα οποία αφορούσαν το τι θα κάνουμε για να ενισχύσουμε το έργο των ομάδων οικονομικών πληροφοριών για να αντιμετωπίσουμε το ξέπλυμα χρήματος και οτιδήποτε αφορά ειδικότερα την τρομοκρατία συμφωνώ με αυτούς, την κυρία Σαρτζεντίνη, την κυρία Γκόμες και άλλους που λένε ότι υπάρχει μια ευρωπαϊκή διάσταση και ότι πρέπει να εστιάσουμε σε αυτόν. Γι' αυτό ακριβώς ε, έκανα και μια ιδιαίτερη προσπάθεια να στηρίξω το έργο που κάνετε στην πέμπτη οδηγία περί ξεπλήματος χρήματος και να υπογραμμίσω ότι αν και όταν, ελπίζω όταν, συμφωνήσατε για την ενίσχυση των μονάδων αυτών και των μητρών διαφάνειας που πάνε πακέτο με τα στοιχεία της τέταρτης και πέμπτης οδηγίας. Κοιτάμε να δούμε το τι μπορούμε να κάνουμε για να τα επεκτείνουμε αυτά. Προφανώς θα το συζητήσουμε μαζί σας, αλλά θα δούμε αν μπορούν οι αρχές αυτές να έχουν πρόσβαση σε εθνικά μητρώα τραπεζικών λογαριασμών και να δούμε πώς θα ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ μονάδων οικονομικών πληροφοριών με τις διοκτικές αρχές για να ενισχυθεί ακριβώς η αρχιτεκτονική σε ένα ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν ξέρω αν σας ενθαρρύνει ή όχι, μπορεί να σας αποθαρρύνει γιατί ε, σημαίνει ότι υπάρχει περισσότερη δουλειά να γίνει. Και βεβαίως ε, συμπάσχω κι εγώ καθώς περνάτε στον ένα το τριμερή διάλογο για τη σχετική οδηγία αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το θέμα γιατί η χρηματοδότηση της τρομοκρατία και το ξέπλυμα χρήματο. δεν πρόκειται να εξαφανιστεί εξελίσσεται και αλλάζει και γίνεται πιο δύσκολο να αντιμετωπιστεί γι' αυτό ακριβώς πρέπει και εμείς να προσαρμόσουμε την δική μας αντίδραση προς την κατεύθυνση των μέτρων που επεξεργάζεστε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι κάλυψα τα περισσότερα. Αν όχι, μπορείτε πάντα να έρθετε σε επαφή μαζί μου Σας ευχαριστώ κύριε Επίτροπε και νομίζω ότι οι συνάδελφοι θα συμφωνήσουν με αυτό το οποίο είπατε. Μιλήσετε για οδηγία ξεπλήματος ε, χρήματος. Ε, καλά, είναι κατά του ξεπλήματος χρήματος, αλλά το ότι έχουμε τον ένα το τριμερή διάλογο που ότι εδώ πέρα δεν είμαστε απλά καφενείο, κάνουμε ουσιαστική δουλειά και βεβαίως ε, είχαμε και αυτή τη συζήτηση γιατί θέλουμε να αναπτύξουμε και στην Επιτροπή μας αυτή την διάσταση της ασφάλειας και οι συνάδελφοι βεβαίως ασχολούνται πάρα πολύ με τις οδηγίες αυτές, ε, αυτήν και τις παρόμοιες με αυτόν τον στρατηγικό στόχο. Και πάλι λοιπόν οι συνάδελφοι έργασαν πάρα πολύ σκληρά για να γίνει αυτό πραγματικότητα. Και να πω επίσης ότι ε, τώρα βεβαίως ε, είμαστε ενεργοί και στην σχετική έκθεση. Αυτή δραστηριοποιούμαστε που θα απασχολεί στην Επιτροπή Τρομοκρατίας και παρακολουθούμε το τι γίνεται και στο Παρίσι, στο Λονδίνο. Σα παρακολουθώ οπωσδήποτε εγώ και ίσω και άλλοι συνάλφοι στο Twitter, αλλά ξέρω ότι είχατε πάει στο Βερολίνο πρόσφατα και κάνετε πολλά και διάφορα. Αλλά είναι ακριβώ η επίσημη επαφή σα με την Επιτροπή μα που είναι πολύ σημαντική. Και είναι σημαντική συζήτηση με ουσία. Σας ευχαριστούμε λοιπόν πάρα πολύ. Ο τρίτος διάλογος ασφαλείας θα είναι στο πρώτο εξάμεινο του 2018 και θέλω η Επιτροπή μας να διατηρήσει ακριβώς αυτή την σχέση με τον διάλογο αυτόν και θα έχουμε μια νέα διάσταση με τα κατόπιν και με την Επιτροπή Περιτρομοκρατίας και στην για την περίπτωση που δεν το ακούσατε αύριο θα παρουσιάσετε το σχέδιο διαλειτουργικότητας και νομίζω ότι θα έχουμε την ευκαιρία να το συζητήσουμε μαζί σας κατόπιν. Νομίζω ότι έχει μεγάλο ενδιαφέρον αυτό και μετά θα είναι μια επιτροπή που θα θα είναι μια έκθεση που που θα θέλει να αναλάβει η επιτροπή μας και θα έχουμε την ευκαιρία να τα συζητήσουμε αυτά μαζί. Σας ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ συνάδελφοι. Ξέρω ότι είναι Δευτέρα βράδυ του Στρασβουργού. Σας ευχαριστώ και πάλι παρόλα αυτά για την ε, συζήτησή μας οι ε, επίτροποι είναι μαθημένοι, δεν αντέχουν. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και την ομάδα σας. Ευχαριστώ συνάδελφοι. Ήταν έξοχη συζήτηση. Μπορούμε να κάνουμε μια διακοπή μέχρι τις 20 και 30 για την ηλεκτρονική ψηφοφορία στις 8.30. Διάλειμμα 5 λεπτών.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 Είμαστε έτοιμοι, συνάδελφοι, ξεκινήσουμε την ψηφοφορία. Αλλά έχουμε κάποια πηγαδάκια για την ψηφοφορία. περιμένουμε να ολοκληρωθούν συζητήσεις. Είναι εδώ η συγκεκριτή. Όταν είστε έτοιμοι και στις θέσεις σας μπορούμε να ξεκινήσουμε. Σε ευχαριστώ Τόμας που με καθησύχασε. Εγώ είμαι έτοιμο, αλλά δεν μου καθίσει όλοι οι συνάδελφοι. Κάποιο δεν έχει κάρτα ψηφοφορία. Η συνάδελφο το είπε, οπότε θα λάβουμε υπόψη την ψήφο τη. Υπάρχει κάποιο άλλο που δεν έχει την κάρτα του. Οπότε ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πολύ μαλακό το σφυράκι. Δεν μου πολύ αρέσει. Συγγνώμη, δεν είναι το συνηθισμένο. Λοιπόν, λοιπόν κατά πολέμηση του ξεπλήματος χρήματος με στο ποινικού δικαίου. Ο Ιγνάθιο Κοράο είναι συγγητής για να ξεκινήσουν θεσμικές διαπραγματεύσεις ε, στην πραγματιστική ομάδα. Πριν ξεκινήσουμε, κατά τμήματα συμφορίε και συμβαστικέ, σύμφωνα το άρθρο 154-5 του εσωτερικού κανονισμού, δεν γίνονται αποδεκτά. Κατά διάρκεια των πραγματεύσεων, μια συμφωνία εξευρέθη μεταξύ συγγητού και σκιωδών και έχουμε συμβασμού 3, 5 και 6 που αυτοί οι συμβιβασμοί πρέπει να είναι ξεχωριστέ ψηφοφορίε στο άρθρο 3, παράγραφος 2α, άρθρο 5, παράγραφος 2α και άρθρο 6, εδάφιο αβ. Λέγοντα αυτά, που καταγράφονται στα πρακτικά. Θέλω να μου πει ο εισηγητή, αν θέλει εν συντομία να πάρει το λόγο, ο κύριος Κοράο. Γρήγορα, γρήγορα. Είμαι ευχαριστημένος που κατάφερα να φτάσω. 15 ώρες ταξίδι. Ευχαριστώ όλους τους εισηγητές, τους χιώδεις εισηγητές με τους οποίους ετοιμάσαμε αυτή την εργασία και καταλήξαμε στην έκθεση. Σημαντικό το έργο για αυτή την Επιτροπή και για το Ευρωκοινοβούλιο. Άλλο ένα βήμα είναι για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. Προσπαθούμε να πλήξουμε τα περιουσιακά του στοιχεία, τα κεφάλαια και κυρίως σε σχέση με την πρόσωπη Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλαμε να καταλήξουμε σε πολιτική θέση πιο προθυμένη από πλευρά Κοινοβουλίου και θέλουμε έτσι να την προωθήσουμε αν καταφέρουμε να, να να πάρουμε την εντολή. Ευχαριστώ εκ νέου όλους τους σκιώδεις ηγητές, όλους όσους συμμετείχαν και κλείνω. Αυτά εντάχει. Ευχαριστώ κύριε Κοράου. Είχαν φρικτά ταξίδια κάποιοι συνάδελφοι προσπαθώντας να έρθουν εδώ. Σας ευχαριστώ που ήρθατε. Ας ψηφίσουμε λοιπόν. Ξεκινάμε από την τροπολογία 28. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβιβασμός που αφορά το άρθρο 1. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβασμός για το άρθρο 2. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 96. Άρχεται η συμφορία. 96. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική το άρθρο 3 πρώτο τμήμα. Άρχεται η συμφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 114 και 115 μαζί. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνονται. Συμβαστική επί άρθρου 4. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Για το άρθρο 5 πρώτο τμήμα. τη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. τη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 144. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 148. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική για το άρθρο 6 άρχεται. Συμφορία πρώτο τμήμα. Για το πρώτο τμήμα. Πέρας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Άρχεται η συμφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 162. Άρχεται η συμφορία. Είναι λίγο αργά τα μηχανήματα. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική για το άρθρο 7. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική για το άρθρο 8. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική το άρθρο 8α νέο. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 173. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική άρθρο 9. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική άρθρο 10. Άρχεται η ψηφοφορία. Α. Συνάδελφοι. Μισό λεπτό. ΔΕΒΕ 28. Άρχεται η ψηφοφορία. Ευχαριστώ που μου το δείξατε, το ξέχασα. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική άρθρο 10. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας εγκρίνεται. Συμβαστική άρθρου 12, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική άρθρου 13, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 30, άρχεται η ψηφοφορία. Στις ιδεολογικές σκέψεις είμαστε τώρα. Πέρας. Εγκρίνεται. 31. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 33. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. εγκρίνεται. Τζούρι 1, άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 34, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Α, απορρίπτεται. Τζούρι 2, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 38. Άρχεται η σοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Οίκον 2. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Τζούρι 3. Άρχεται η Πέρας. Εγκρίνεται. ΔΕΒΕ 2 και τροπολογία 1 ταυτόσημες άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνονται. Τροπολογία 41 άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 42 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Ή 3 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 43 άρχεται η ψηφοφορία. Συγγνώμη λέει ο πρόεδρος. 46 άρχεται η ψηφοφορία. Τροπολογία 46. Πέρας. απορρίπτεται. Τζούρι 4 άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Δεβε 3 άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Τεπολογία 47 ξεκινάμε. Τέλος. Απορρίπτεται. Τροπολογία 48. Ξεκινάει η ψηφοφορία. Τέλος. Απορρίπτεται. Τζούρι 5. Ξεκινάμε. Τέλος. Εγκρίνεται. Τροπολογία 50. Ξεκινάμε. Τέλος. Α, απορρίπτεται. Τροπολογία 52, πρώτο τμήμα. Ψηφίζουμε. Τέλος. Α, απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα. Ψηφίζουμε. Τέλος. Α, απορρίπτεται. Τροπολογία 57. Ψηφίζουμε. Τέλος. Απορρίπτεται. Τζούρι 7. Ψηφίζουμε. Τέλος. Εγκρίνεται. Τοπολογία 58. Ψηφίζουμε. Τέλος. Εγκρίνεται. Τροπολογία 63. Ξεκινάμε. Τέλος. Απορρίπτεται. Τροπολογία 64, πρώτο τμήμα, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα. Ξεκινάμε. Πέρας. Απορρίπτεται. ΔΒ5. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. εγκρίνεται. Τροπολογία 65. Ξεκινάμε. Τέλος. Απορρίπτεται. 66. Ξεκινάμε. Τέλος. Εγκρίνεται. Οίκον 6. Ψηφίζουμε. Εγκρίνεται. ΔΕΒΕ 6. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Τοπολογία 74. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Dev 7. Ψηφίζουμε. Τέλος. Απορρίπτεται. Τζούρι 14. Ψηφίζουμε. Τέλος. Εγκρίνεται. Τροπολογία 73. Άρχεται η ψηφοφορία. Συγγνώμη, ο Πρόεδρος. Τροπολογία 73 μέχρι 75 μέχρι 85 όλο μαζί. Ξεκινάμε. Τέλος. Απορρίπτονται. Ψηφίζουμε την τζούρι 12. Τέλος. Εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία, μονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται. Πέρας. 39 ψήφοι υπέρ, καμία ψήφος κατά και τέσσερις αποχές για την έναξη διαπραγματεύσεων. Απόφαση για να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις άρχεται. Πέρας. Κάποιος δεν ψήφισε. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται 38 ψήφοι υπέρ, καμία ψήφο εναντίον και δύο αποχέ. Συγχαρητήρια λοιπόν στον εισηγητή και στους κοιόδης εισηγητές. Ευχαριστώ συνάδελφοι. Κάποιοι συνάδελφοι πέρασαν πολύ δύσκολο ταξίδι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τελειώσαμε τις ψηφοφορίες. Είναι και η τελευταία συνεδρίαση του έτους. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνεργασία σας. Ευχαριστώ τους κλητήρες. Καλά Χριστούγεννα. Στεπανιδή. Τα λέμε